Η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα στις 12 η ώρα. Επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης ε, η ερώτηση προς την Κομισιόν που αφορά την επιδημία Schmallenberg. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο καταρχήν ε, σε αυτούς ε, που συνέταξαν την προφορική ερώτηση. Αρχίζει ο κύριος Λεγιαρίκ για δύο λεπτά παρακαλώ. μετά από την ε, τρελή αγελάδα, τη φυματίωση, τον καταρροϊκό πυρετό, τον αυθόδη πυρετό, έχουμε τον νέο ιό, τον ιό Σμάλεμπερκ που πλήττει τις εκτροφές μας και τα αποτελέσματα ε, δεν θα φανούν λίγες ε, εβδομάδες. Θα γίνει σφαγή βοηδών και θα ήθελα να ρωτήσω, κυρία Επίτροπε, τι μπορείτε να κάνετε έτσι ώστε να μην τεθεί εμπάργο στο βόλιο κρέας μας. Μπορούμε να ανοιχνεύσουμε καλύτερα αυτή την ασθένεια και να την περιορίσουμε. Επίσης θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό ταμείο αποζημιώσεων, σε συνεργασία με σε συνεργασία με κράτη-μέλη. Αυτή η, ε, υγειονομική κρίση δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε κινδύνους και να διακυβεύσει τις ελεύθερες συναλλαγές. Επίσης δεν θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την διατροφική αλυσίδα. Όλα αυτά δεν θα πρέπει να μας απασχολήσουν μέσα στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο Λεγιαρίκ. Ακολουθεί ο συνάδελφο Νίκολσον για δύο λεπτά παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρο. Είναι ατυχέ που εμφανίστηκε η ασθένεια Σμάλενμπεργκ διότι οι επιπτώσει είναι σημαντικέ σε αυτή τη φάση ε, του χρόνου Είχαμε κάποιες περιπτώσεις του φθονόπορου αλλά τώρα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Ε, γεννούνται πολλά νεκρά από τα παιδιά και νομίζω ότι πρέπει να παρατρύνουμε μία αναλογική ανταπόκριση. Ο, θεωρείται ότι ο ιός δεν είναι επιθετικός για τον άνθρωπο και γι' αυτό δεν Πιστεύω ότι η απαγόρευση εισαγωγών κρέατος ας πούμε και γάλακτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Αίγυπτο και από τη Ρωσία είναι υπερβολικά. Η μετάδοση του ιού μπορεί να προκαλέσει βεβαίως διασυνοριακά προβλήματα. Είναι αδύνατο να ελέγξουμε τη μη μεταφορά του τις περισσότερες φορές. Χρειαζόμαστε μια συντονισμένη ανταπόκριση από τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να διαδώσουμε τα στοιχεία για να αποκτήσουμε μια αληθινή εικόνα της επέκτασης του ιού. Μέτρα πρέπει να ληφθούν για να καθησυχάσουμε τους συνεταίρους μας όσον αφορά την υψηλή ασφάλεια των τροφίμων της Ευρώπης. Χρειάζεται ακόμη να επινοηθεί για κάποιος εμβολιασμός μελλοντικά ώστε η γεωργία να την Ευρώπη να μην έχουν να αντιμετωπίσουν τέτοια κατάσταση μελλοντικά. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο Νίκολσον. Ο συνάδελφος κύριος Ντες έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συζήτηση για τις ασθένειες ε, των ζώων, ε, η ασθένεια που προκαλείται από τον ιό Σμάλενμπεργκ. Οι επιστήμονες έχουν αποφανθεί, ο ιός αυτός ε, μοιάζει με τον ιό Ακαπάνη που εμφανίζεται και πλήττει ζώα από την Αφρική μέχρι την Αυστραλία. Ο ιός Ακαπάνη είναι ακίνδυνος για ανθρώπους που σημαίνει μπορούμε να θεωρήσουμε ότι και ο ιός Σμάλενμπεργκ είναι ακίνδυνος για τους ανθρώπους. Όμως ε, είναι μεγάλος κινδύνος για τα ζώα και προκαλεί πολλές ζημιές. Κυρία Επίτροπε, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιοριστεί αυτή η ασθένεια. Ε, πρέπει να αναλυφθούν αποτελεσματικά μέτρα και έτσι λοιπόν ε, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση θανάτωσης ακριβώς όπως έχει συμφωνηθεί στη Γερμανία. Ο ιός αυτός όπως ακούστηκε μεταφέρεται από κουνούπια και νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί προστασία. Η προστασία βέβαια μπορεί να υπάρξει μόνο από εμβόλιο και εκ μέρους της ΕΛΚ καλούμε εμεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να ε, υποβοηθήσει την παραγωγή εμβολίου, να διατίθεται αυτό στο εμπόριο. Και είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να ε, επεξεργαστεί τα απαραίτητα στοιχεία για να μπορούν και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Εκτός αυτού είναι και καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να υπάρχουν εμπορικοί περιορισμοί όπως ε, προβλέπεται στις 23 Εν τω μεταξύ βέβαια ε, μπορούν και ίσως και αυτοί να έρθουν Ρωσία, Αίγυπτος, Ηνωμένε Πολιτείε έχουν επιβάλει περιορισμούς και όσο ταχύτερα αντιδράσουμε, ε, τόσο περισσότερο περισσότεροι τότε υπάρχουν να μην επεκτατεί η ασθένεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ντές. Ο κυρία Μπρίτα Ράιμερς ε, για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Στη διάρκεια του τελευταίου έτους ε, διαπιστώσαμε αυτή τη νέα ασθένεια η οποία από ό,τι φαίνεται ε, μεταδίδεται μέσω των εντόμων και δημιουργεί ε, δυσμορφίες κυρίως στα εγωπρόβατα. Υπάρχουν μια σειρά από ζημίες για τους παραγωγούς που μέχρι τώρα έχουν μείνει αβοήθητη. Θα πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε επί τη βάση επιστημονικών δεδομένων να προσπαθήσουμε να δούμε κατά πόσο πρόκειται για ένα νέο ιό ή όχι. Χρειάζεται χρόνος βέβαια, ενώ στην πραγματικότητα μας λείπει ο χρόνος, διότι πρέπει να υπάρχουν κατάλληλη βοήθεια. Θα μπορούσε ίσως να υπάρχει κάποιο ταμείο. Θα πρέπει όμως να γίνονται κατάλληλε κοινοποίησει ακόμα και αν υπάρχει ταμείο. Όταν Πότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να εκπονήσει μια νέα ε, μεθοδολογία για τις ασθένειες ε, ώστε να μπορεί να παράσχει και ενισχύσεις αλλά και δυνατότητες παρακολούθησης για όσους ε, πλήττονται από αντίστοιχες ασθένειες. Υπάρχει ελάχιστος χρόνος ε, η ασθένεια μεταδίδεται και ε, μειώνονται οι εξαγωγές ε, από τις τρίτες χώρες. Υπάρχουν λοιπόν συνέπειες για όλους τους κτηνοτρόφους και παρά το γεγονός ότι μεταδίδεται μέσω εντόμων υπάρχουν ελάχιστες δυνατότητες να ελέγξουμε την κατάσταση. Ε, πώς σκοπεύει λοιπόν να δράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν μια σειρά από ασθένειε, οι οποίες ε, εισάγονται σε κάποιες περιπτώσεις αλλά επειδή ακριβώ αυξάνεται και η μεταφορά ζώων ε, μπορεί και να μεταδίδονται πολύ περισσότερο. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για όσους ε, πλήττονται από την ασθένεια, γεγονό που θα βοηθήσει όλου μα. Η κυρία ε, Χέντεγκαρτ, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Ντάλι δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Θα απαντήσω λοιπόν εγώ στις ερωτήσεις σα εκ μέρου τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρακολουθήσει την εξέλιξη του θέματος αυτού του Σμάλενμπεργκ ευθύ εξ αρχή και εξακολουθούμε να συντονίζουμε την ευρωπαϊκή απάντηση. Να πω ήδη ευθύ εξ αρχή στην κυρία Ράιμέρ, ότι υπάρχει μία ε, διαδικασία την οποία ακολουθούμε συνήθως για νέες νόσους. Ε, υπάρχουν μηχανισμοί για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει κατάλληλη απάντηση σε οποιαδήποτε επιδημία και αυτό μας επιτρέπει να εντοπίσουμε τον ιό και να ετοιμάσουμε συντονισμένες δράσεις. Οι πρόσφατες εξελίξεις όπως για παράδειγμα η απάντηση στο ΙΤΑ 1 ε, καταδεικνύει ότι το επίπεδο προετοιμασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ικανοποιητικό και ε, η επαρκής πρόληψη οδηγεί σε κατάλληλες αντιδράσεις. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ρυθμίσουμε σε κάποιες περιπτώσεις τους υφιστάμενους μηχανισμούς και στη νέα στρατηγική για την υγεία των ζώων λαμβάνονται και περαιτέρω δράσεις προκειμένου το επίπεδο προετοιμασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βελτιωθεί περαιτέρω. Υπάρχει και ένα έγγραφο καθοδήγηση το οποίο αναφέρει τι βασικέ δράσει που πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το έχει ετοιμάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το έχουν εγκρίνει εμπειρογνώμονε και ενδιαφερόμενοι στα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τώρα την πρόληψη τη περαιτέρω εξάπλωση του ιού, ε, παρά το γεγονό ότι ο ιό αυτό έχει ήδη μεταδοθεί ε, σε οκτώ κράτη-μέλη ε, στα ζώα των κρατών μελών, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει απειλή για την περαιτέρω εξάπλωση στη διάρκεια της ε, τρέχουσα εποχής. Πρέπει αυτή τη στιγμή να επαγρυπνούμε, αλλά αυτό ούτω ή άλλω το κάνουμε. Θα πρέπει να σας πω ότι η εξαγωγή ε, άρρωστων ζώων δεν επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποια μέτρα λάβουμε θα πρέπει να είναι αναλογικά και βιώσιμα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες υποδηλώνουν ότι οι επιπτώσεις αυτής της νόσου για την υγεία των ζώων και την αναπαραγωγή είναι περιορισμένες και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα μπορούσε να προκαλέσει ασθένεια και σε ανθρώπους. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την ε, ΕΦΣΑ, την Ευρωπαϊκή Αρχή για Τρόφιμα, να συλλέξει ε, στοιχεία για να δει τι συνέπειες υπάρχουν στην υγεία των ζώων και την αναπαραγωγή τους για την επιδημία της ε, Σμάλεμπερ, καθώς επίσης και για την ευημερία των ζώων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται σε επαφή με τα κράτη-μέλη ε, για να ε, μαζέψει δεδομένα και από εκεί και πέρα μετά τη συλλογή των δεδομένων αυτά θα διαβιβάζονται στα κράτη-μέλη. Ε, ε, το κενό που υπάρχει αφορά το γεγονός ότι αυτή η νόσος είναι νέα. Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το κενό ε, έχουμε ζητήσει μελέτες ε, για να έχουμε μία ε, συγκεκριμένη κτηνιατρική πολιτική και μπορεί να ληφθούν και άλλα προληπτικά μέτρα ελέγχου είτε σε επίπεδο κρατών μελών είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως γίνεται και με τις υπόλοιπες ιογενείς νόσους, δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία για θεραπεία των ζώων που έχουν επληχθεί από την νόσο από τον ιό του Σμάλενμπερ και δεν ξέρουμε πότε θα είναι έτοιμο και το εμβόλιο όσον αφορά τους πιθανούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία από τον ιό αυτό, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Ασθενειών και Ελέγχου δήλωσε πέρσι ότι δεν υπάρχει πιθανότητα αυτός ο νέος ιός να μεταδοθεί και στους ανθρώπους και τα τρέχοντα στατιστικά δεδομένα υποστηρίζουν αυτή την αξιολόγηση. Ωστόσο, δεν μπορούμε τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο να το αποκλείσουμε. Εάν υπάρξουν νέε ενδείξει ε, ότι μπορεί να υπάρχει κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα, θα ζητήσει συγγνώμη, από την ε, Υπηρεσία Πρόληψη και Ελέγχου να μα δώσει μια επικαιροποίηση και να δούμε τι μέτρα μπορούμε να λάβουμε. Θα προσπαθήσουμε να ε, αντιδράσουμε ε, μέσω του συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταχείας αντίδρασης. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η αυστηρή προσέγγιση, ε, ένα τρίτο των χωρών έχουν κάνει αίτηση ή σκοπεύουν να κάνουν αίτηση για μέτρα πρόληψης που σχετίζονται ε, με τον ιό αυτό και τις εξαγωγές. Ε, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Νόγκορσον που ζήτησε να έχουμε μια αναλογική απάντηση και ε, θέλουμε να έχουμε και περιοριστικά μέτρα κατά της εξαγωγής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να ζητήσουμε να μην είναι δυσαλάλογα και να υπάρχει αιτιολόγηση μέσω επιστημονικών δεδομένων. Ζητάμε συνεργασία με τρίτες χώρες για να προλάβουμε και να μειώσουμε τους περιορισμούς που έχουν επιβάλει στο εμπόριο. Ολοκληρώνοντα, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη μια αναλογική απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μην υπάρχουν στρεβλώσει τη αγορά και στην εσωτερική αγορά και στο εμπόριο με του διεθνεί μα εταίρου. Θεωρούμε ότι είναι υψή τη σημασία να ε, συνεχίσουμε να έχουμε τα θέματα αυτά υπό τη δέουσα προοπτική. Ευχαριστώ κυρία Χέντεγκαρτ και τώρα ακολουθούν οι ομιλητέ εν ονόματι των πολιτικών ομάδων και καταρχά η κυρία Ντελάνια για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ ο, κύριε Πρόεδρε. Όντως άκουσα την ε, Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή να λέει ότι θα κάνει εποπτεία, θα κάνει μελέτες αλλά χρειαζόμαστε δράση δράση ε, και για τις αγορές και για τους πολίτες οι οποίοι ανησυχούν για την υγεία τους. Όταν λοιπόν κοιτάξω τις αγορές που έχουν κλείσει για τα για τα ζωικά προϊόντα βλέπουμε ότι δεν έχουν κλείσει μόνο για τα ζωντανά ζώα αλλά και για ζωικά προϊόντα και υπάρχουν διαφορετικές προϋποθέσεις για να άρουν αυτές τις, αυτά τα μέτρα. Πάντοτε λοιπόν λέγεται ότι πρέπει να υπάρχει αποκλειστική αρμοδιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι διμερείς ε, συνεννοήσεις αλλά όσο πιστεύουν ότι ε, μπορούν ε, οι χώρες να επιτύχουν κάτι καλύτερο και πιο γρήγορα μόνες τους θα προσπαθήσουν να έχουν μία λύση. Θα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν ενιαία πιστοποιητικά, ενιαίες λύσεις. Χαίρομαι ότι λέτε ότι δεν είναι κάποιος ιός που μπορεί να μεταφερθεί στον άνθρωπο αλλά θα πρέπει να το λέτε πιο ευκρινό στην ανακοίνωσή σας για να κάνει Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκρότε τώρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για τη δυνατότητα η οποία δίνεται τώρα να συζητήσουμε το θέμα αυτό μεταξύ μας στη χώρα μου στην Δυτική Γερμανία υπάρχουν 900 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί και υπάρχει και μία συζήτηση στο κοινό. Υπάρχει ένας φόβος σχετικά με την κτηνοτροφία. Υπάρχουν σημαντικές ζημίες αλλά και θέματα υγείας. Δεν μπορεί κανείς αυτή τη στιγμή να αποκλείσει 100% ότι ο ιός αυτός δεν θα μεταδοθεί στον άνθρωπο και η ΕΦΣΑ ήδη είπε ότι με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Προλήψεως και Ελέγχου συνεργάζεται στενά κατά τρόπον ώστε να μπορέσει να παρακολουθεί την ε, υγεία και για τους ανθρώπους ε, και υπάρχει μια διαδικασία ε, εποπτείας έχει γίνει και μια προσωμείωση και ελέγχθη ότι 8 κράτη είναι, έχουν ήδη από αυτό τον ιό και βλέπουμε ότι την άνοιξη και το καλοκαίρι με τις ε, μύγες θα επεκταθούν αυτοί οι έχουν διαγραφεί διάφορα σενάρια. Μπορεί λοιπόν να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τι μέτρα σκοπεύει να λάβει ή λαμβάνει ήδη για να καταπολεμήσει τους κινδύνους που διαγράφησαν στην προσωμείωση. Έχει γίνει μία λεπτομερής ανάλυση διότι καλό θα είναι να εντοπιστεί και να παρεμποδιστεί ο ιός αυτός διότι ε, πρέπει να βρεθούν μέτρα για να καλαπολεμήσουμε τελεσίδικα αυτό το μέτρο αλλά ε, τι έχει ληφθεί κατά τρόπον ώστε να μην, ε, να μην επεκταστεί ο ιός και στα 27 κράτη προς το παρόν ή έχει, βρίσκεται στα 8 αλλά δεν πρέπει να παρέμβει τα υπόλοιπα σύνορα. Ευχαριστώ κύριε Γκρότε. Ο κύριος Έλγουαρτ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην Ιρλανδία δεν έχει αναφερθεί κρούσμα του ιού Σμάλεμπεργκ. Ελπίζουμε να μην γίνει ούτε στο μέλλον κάτι αντίστοιχο. Πάντως με ανησυχεί τι γίνεται ε, με τις αποστολές ε, από Ρωσία, Κίνα και άλλες χώρες τέτοιων ε, ζώνων 20 Μαρτίου και μετά. ίσως γίνουν ε, εισαγωγές ε, από τις χώρες αυτές και, σε άλλα, και από άλλα ε, ζώα. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και το χείριο κρέας. Πρέπει να λάβουμε δράση άμεσα για να προστατεύσουμε τη φήμη των ευρωπαϊκών προϊόντων. Και χαιρετίζω την πρόταση της Κομισιόν να μην δεχτεί την επιβολή περιορισμών από τρίτες χώρες. Θα πρέπει πάντως να κάνουμε προσπάθειες να μην πέσει η κτηνοτροφία μας σε θύμα αυτής της κατάστασης. Πρέπει σε όλους τους καταναλωτές και εμπορικούς εταίρους να τους ενημερώνουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χόισλινγκ για ένα λεπτό. Ναι, η χθεσινή αριθμή είναι σαφής. Βλέπουμε ότι πέραν των 900 ε, ε, επιχειρήσεων έχουν πληγεί στη Γερμανία και 8 χώρες στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όταν λοιπόν επεκταθεί ε, σε ολόκληρη την Ευρώπη ο ιός αυτός θα έχουν μείνει μόνοι τους οι γεωργοί, δεν θα υπάρχει καμία αποζημίωση γι' αυτό και είναι ακατανόητο για μένα γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να μειώσει τη σημασία του πριών του προβλήματος αυτού. Χρειαζόμαστε την εμπλοκή των ε, επιστημόνων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και πρέπει να βοηθήσουμε και τους ε, ε, κτηνοτρόφους που έχουν εγωπρόβατα. Ήδη είχαν πληγεί από τον αυθόδη πυρετό και τον καταραϊκό πυρετό και τώρα δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν όλες αυτές οι ασθένειες οι οποίες οφείλονται στις κλιματολογικές κλιματολογικές αλλαγές, γι' αυτό και πρέπει να καταπολεμήσουμε τις κλιματολογικές αλλαγές. Ευχαριστώ τον κύριο Χόισλινγκ. Ε, η κυρία Γκίλινγκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από ό,τι καταλαβαίνω πρόκειται για έναν νέο ιό. Εδώ και δύο δεκαετίες δεν είχαμε ξαναδεί έναν καινούριο ε, ιό. Στη δική μας περιφέρεια γραμμικά 200 μίλια από βορρά προς νότον έχει ανιχνευτεί η παρουσία του ιού και εξαπλώνεται ταχύτατα. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση συγκεκριμένα. Πρώτα απ' όλα να αναγνωρίσετε τη σημασία της ανάληψης ταχείας και αποφασιστικής δράσης. Δεύτερον, τι εμπορικοί ε, περιορισμοί και τι επιπτώσεις θα υπάρχουν. Αυτό πρέπει να το δείτε. Επίσης, έρευνα, ταχεία έρευνα για πιθανό εμβολιασμό και αντιμετώπιση. Να συγκεντρωθούν επίση αξιόπιστα δεδομένα. Και τέλο, αν είναι δυνατό, γιατί είναι κατά την άποψή μου το σημαντικότερο, αυτό να το αντιμετωπίσετε ω προειδοποίηση. Σίγουρα αλλάζουν και τα κλιματικά πράγματα, οι κλιματικέ ε, συνθήκε και αν αρχίσει να ε, μπαίνει στο σύστημα και στην τροφική αλυσίδα μια ολόκληρη σειρά από ιούς θα το να το αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ κυρία Γκίρλινγκ. Τώρα υπάρχουν οι άλλοι εγγεγραμμένοι ομιλητές και ξεκινά ο κύριο Νικολέσκου για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Δύο πτυχέ ε, έχει συζήτηση κατά την άποψή μου. Πρώτα απ' όλα τη σοβαρότητα. Πρέπει να δούμε πόσο σοβαρή είναι αυτή η επιδημία. Ξεκίνησε πριν από πέντε μήνε, αλλά ο ιό προπήρχε σε τουλάχιστον 1.200 γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν έχουμε ακόμη ε, την κατάλληλη ενημέρωση. Είναι ε, οι πληροφορίες λίγο κατακαιρματισμένες. Δεύτερον, ποιες είναι οι επιπτώσεις για τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Πρέπει να δούμε και την κατάσταση των ζώων, αλλά και τους περιορισμούς στις εξαγωγές που έχουμε βάλει στους εταίρους μας. Οι εμπορικοί περιορισμοί δεν δικαιολογούνται, είχατε πει σε απάντησή μας, ε, σε απάντηση ε, σε ερώτησή μας τον Ιανουάριο. Ε, τώρα οι εισαγωγές από τα κράτη-μέλη αξιολογούνται, ε, θα αξιολογηθούν μάλλον από τις 20 Μαρτίου και οι εκτινοτροφικές οργανώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνουν στη Ρωσία πληροφορίες για την καταπολέμηση του και στη Ρωσία. Θα πρέπει όμως να μας δώσει η Κομισιόν πιο πολλές πληροφορίες ό,τι αφορά ε, τους Ρώσους. Τι κάνουν οι Ρώσοι, τι ενημέρωση δίνουν ε, στις κτηνοτροφικέ οργανώσεις. Να δούμε και τι έχει γίνει κατά το παρελθόν ε, από πλευρά συμβατότητα των ε, λαμβανών μέτρων με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Θα έχετε διάλογο με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Πώς προτίθεστε να προχωρήσετε. Ευχαριστώ κύριε Νικολέσκου. Τώρα για δύο λεπτά η κυρία Ρόντουστ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Χαιρετίζω το γεγονός ότι υπάρχει σήμερα αυτή η προφορική ερώτηση σχετικά με ε, τον ιό Σμάλενμπερκ και μας ε, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις ε, ιώδεις ασθένειες διότι στην Γερμανία έχουν πληγεί 944 επιχειρήσεις από αυτόν τον ιό και δημιουργούν δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα. Στο Σλέζιβι Χολστάιν στην περιοχή μας επειδή υπάρχει εγκύτητα στις ακτές υπάρχουν πολλά εγωπρόβατα και έχουν πληγεί ο ιός αυτός για πολλές επιχειρήσεις αποτελεί ένα κίνδυνο για εξόντωση και υπάρχουν πάρα πολλά εγωπρόβατα αλλά και βοήθεια που έχουν πληγεί από τον ιό αυτό και τους τελευταίου, τις τελευταίες εβδομάδες ε, από 106 ε, αυξήθηκαν σε 116 οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μολυνθεί με τον ιό αυτό και ε, με τα θνησιγενή νεογνά πλήττονται διπλά οι επιχειρήσεις. Θέλω λοιπόν να ότι δεν είναι δυνατόν, χρειαζόμαστε ένα εμβόλιο επιγόντων. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω αν έχει προχωρήσει η έρευνα και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τις επιχειρήσεις ε, στην έρευνα για να βρεθεί ένα τέτοιο εμβόλιο. Επίσης πρέπει να δούμε αν ε, μπορούν να αποζημιωθούν και να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποστεί σωμαρές οικονομικές ε, ζημίες λόγω του ιού αυτού. Παρακαλώ δράστε γρήγορα και κρατήστε μας συνεχώς ενημέρους για το τι γίνεται διότι οι γεωργοί προσβλέπουν προς εσάς αλλά και προς εμάς. Ευχαριστώ κυρία Ρόντους. Τώρα για 1,5 λεπτό ο κύριος Σνέλχαρτ. Κυρίες και κύριοι, κυρία Επίτροπη, βέβαια είναι σωστό ότι σήμερα μιλάμε στο Κοινοβούλιο για τον ιό Σμάλενμπεργκ. Θα θέλω όμως να παρακαλέσω να μην πανικοβαλόμαστε και να είμαστε πιο ήρεμοι, διότι πολλές, ε, όπως και στο παρελθόν, έχουμε συναντήσει αυτόν τον ιό, όπως και στο παρελθόν, βέβαια σε μεγαλύτερους αριθμούς μολύνσεων και βλέπουμε ότι τα ζώα μπορούν μόνοι τους να δημιουργήσουν ανοσοποιητικό σύστημα για κατά αυτής της Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν για την γρήπη των πτηνών. Είχαμε λάβει πάρα πολλά μέτρα και μετά έπρεπε ε, να υπεραμεινθούμε και να δικαιολογηθούμε διότι οι πράσινοι μας επέπληξαν ότι υπήρξαν χρεοκοπίες και ότι είχαμε ε, υπερβάλλει. Βέβαια πρέπει να ληφθούν μέτρα, πρέπει να δούμε πόσα και τι μέτρα χρειάζονται αυτή τη στιγμή αλλά ζητάμε αμέσως αποζημιώσεις νομίζω ότι είναι παρατραβηγμένο. Υπάρχουν οι δυνατότητες στην στην ε, Γερμανία, στην Ολλανδία να υπάρξουν επεμβάσεις και θα παρακαλούσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να ε, στηρίξει την εθνική λύση για το πρόβλημα αυτό αντί να επέμβει κατευθείαν η Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σνέλχαρτ και τώρα ερχόμαστε στη διαδικασία Catch the Eye και καταρχήν δίνω το λόγο στον κύριο Γιάρ για ένα λεπτό. Θεωρώ ότι είναι σωστό να συζητάμε αυτό το πρόβλημα σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τουλάχιστον τρεις πτυχές υπάρχουν στο πρόβλημα αυτό. Καταρχήν ε, οι ε, κτηνοτρόφοι που έχουν πληγεί γιατί όπως ελέγχει όσοι έχουν ε, εγωπρόβατα και πολύ χαμηλή αποδοτικότητα έχουν πληγεί περισσότερο σε ορισμένες ε, περιοχές και θα έπρεπε να εφαρμοστεί η αρχή της επικορικότητος, να υπάρχει διευκρίνηση αλλά και μία αποτελεσματική επέμβαση. Υπάρχουν βέβαια μία δεύτερη πτυχή των καταναλωτών οι οποίοι πρέπει να ενημερωθούν διότι βλέπουμε ότι ε, καθημερινά ε, θα πρέπει να ενημερώνονται να ξέρουν αν ο ιός αυτός είναι επικίνδυνος ή όχι. Όχι μόνο με επιστημονικές δηλώσεις ακατανόητες. Και τρίτον, χρειάζεται ανάλυση και έρευνα η οποία θα πρέπει να συντονιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ κύριε Γιάρ. Ο κύριος Όμπερ Μάιερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάνω από χίλιες ε, επιχειρήσεις έχουν πληγεί από τον ε, ιό αυτό και ε, με την αύξηση της θερμοκρασίας στην άνοιξη θα αυξηθεί ο αριθμός και των πληγέντων επιχειρήσεων. Αλλά σε χώρες όπως στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στην Αγγλία παρουσιάζονται και νέες μολύνσεις, νέες ασθένειες και πρέπει να δούμε ε, πώς αυτό ε, εμπλέκει και τους ανθρώπους και θυμάστε ότι είχαμε στην Αυστρία τέτοια προβλήματα και γι' αυτό πιστεύω ότι καλύτερο είναι να προλαμβαίνουμε ε, και αντί όπως τώρα να πρέπει να κάνουμε να λαμβάνουμε επίγοντα μέτρα για να μπορέσουμε να πατάξουμε τις πολύ επίγουσες καταστάσεις. Ευχαριστώ Παρακαλώ να σας πω ότι δεν επιτρέπεται να χειροκροτείτε στο Κοινοβούλιο και ανεφέρομαι στα ανώτερα έδρανα. Και τώρα έχει τον λόγο η κυρία Χέντεγκραου. Ευχαριστώ. Αυτή η απειλή αποτελεί έναν ακόμα λόγο για να αναπτύξει ε, πρότυπα ε, ζωικής υγείας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς ε, το εμβόλιο για τον ιό ακόμα είναι στη φάση προετοιμασίας και η επιδημία θα έχει σοβαρές επιπτώσεις ιδίως κατά τη διάρκεια του μηνός Απριλίου. Επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να δίνονται πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ε, στα κράτη-μέλη. Επίσης θα πρέπει να προστατεύσουμε τις περιοχές οι οποίες ακόμα δεν έχουν πληχθεί από τον ιό για να εξετάσουμε ε, τους διαδρόμους ε, μετάδοσης. Πρέπει να υπάρχει σωστή διάγνωση και να ενημερώνονται οι εθνικές αρχές για τα διάφορα κρούσματα ώστε να απομονώνονται οι αιστείε θα πρέπει, ε, όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα πρόορης διάγνωσης. Πώς σκοπεύετε να ενημερώσετε τους κτηνοτρόφους στις περιοχές που έχουν ε, κρούσματα του ιού. Ευχαριστώ την κυρία Μπασέσχο. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία Catch the Eye και δίνω το λόγο στην Επίτροπο κυρία Χέντεγκαρτ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα για τον κύριο Χόσλινγκ να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παραγνωρίζει την σημασία του προβλήματος για την κυρία Γκέρλινγκ, η οποία ανέφερε κάποια πράγματα που θα μπορούσε να πράξει η Κομισιόν, εμπορικές πτυχές, συγκέντρωση δεδομένων κλπ. κλπ. Νομίζω ότι αναφέρθηκα σε όλα αυτά και είπα ότι εντάσσονται στη δράση που έχουμε ήδη αναλάβει. Σε ό,τι αφορά τώρα την κυρία Ντελάνγκη και άλλους που ανησυχούν για τις 10 χώρες που έχουν απειλήσει να επιβάλλουν εμπορικούς περιορισμούς, Θέλω να απαντήσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε επικοινωνία και έχει διάλογο με τις χώρες αυτές. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο Επίτροπος ε, Ντάλι έχει επαφέ με τις ρωσικές αρχές και αυτή τη στιγμή υπάρχει αντιπροσωπεία της Κομισιόν στη, Μοσκού, στη Μόσχα, συγγνώμη, η οποία ακριβώ ασχολείται με το ζήτημα αυτό. Για να ολοκληρώσω λοιπόν, όταν ε, νέε ε, νόσοι, νέοι κίνδυνοι ανακύπτουν, τι κάνουμε, συντονίζουμε τις προσπάθειές μας, ανταλλάσσουμε δεδομένα, ε, συμβουλευόμαστε επιστημονικούς φορείς για να συλλέξουμε στο δυνατόν περισσότερες γνώσεις και ένα από τα μέρη που μπορεί κανείς να βρει επικαιροποιημένε πληροφορίες είναι αυτό το έγγραφο καθοδήγησης ε, στην ιστοσελίδα μας, το οποίο εύκολα επικαιροποιείται όταν προκύψουν νέα δεδομένα, νέες γνώσεις ή ε, λάβουμε στη διάθεση μας περαιτέρω πληροφορίες. οι ενώσει των αγροτών και τα κράτη-μέλη έχουν συμφωνήσει να βρίσκεται, να είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα αυτό το guidance document, το έγγραφο καθοδήγηση και μπορείτε να το συμβουλευτείτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Με συγχωρείτε που υπάρχει τέτοια βοή μέσα στην αίθουσα. Ε, θα μπορούσαμε να κάνουμε και μεγαλύτερο διάλειμμα αλλά δεν είναι πολύ πειθαρχημένοι οι συνάδελφοι και βλέπω ότι υπάρχουν τουλάχιστον πέντε συνάδελφοι οι οποίοι είχαν λάβει το λόγο. Τώρα όμως θα διακόψουμε μέχρι τις ψηφοφορίες πληροφορίες της συνεδρίασης.